πολύ καλό το ότι σήμερα λέμε ότι το ψήφισμα δεν αφορά συγκεκριμένο κόμμα, αφορά τους Ουκρανούς όλους. Και το υφετήσαμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ κύριε Κόβαλ. Ακολουθεί για ένα λεπτό από την ομάδα της Νομόσπονδης Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Βόρειας Καναδική Αριστερά, ο κ. Κόολιτσεκ. Ευχαριστώ. Ε,